Good morning everybody. Sorry for being a little bit late. Καλημέρα σας. Ε, συγγνώμη που καθυστέρησα λίγο, αλλά υποδέχτηκα μία ομάδα εκτός του κτηρίου να περάσουμε στην ε, έγκριση της ημερησίας διάταξης. Παρατηρήσεις, δεν βλέπω. Ανακοινώσεις του Προέδρου, σημείο 2, δεν έχω ανακοινώσεις. Πάμε λοιπόν κατευθείαν στο σημείο 3, πλαίσιο για την ανάκαμψη και εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλωμένων. Οι εισηγητές μας είναι και η Σβίνμπουρν και Γιάκοπ Φον Βάιστσάκερ. Καταρχήν οι κυρίες, παρακαλώ. Και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντα όλου του συναδέλφου για τι τροπολογίε που κατέθεσαν. Νομίζω ότι έχουμε περίπου 400 τροπολογίε που έχουν κατατεθεί και θα επικεντρωθώ σε κάποια κυρία σημεία που είχαμε εντοπίσει ήδη ως συνεισηγητές. Έτσι λοιπόν θα αναφερθώ στις τροπολογίες ανάλογα με τα θέματα που καλύπτουν. Ε, ε εμείς οι ίδιοι είχαμε ως συνεισηγητές καταθέσει περίπου 100 τροπολογίες και προσθέσαμε κάποιο χρώμα στο αρχικό κείμενο. Είμαι ικανοποιημένη που βλέπω ότι αυτά τα κοινά θέματα προέκυψαν επίσης ε, Παραδείγματο χάρη, η περιορισμένη χρήση των δημοσίων πόρων είναι σημαντικό αυτό να γίνεται σε έσχατη ε, λύση, ως έσχατη λύση. Επίσης, οι διασφαλίσει για του πελάτε είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα και χαίρομαι που και οι υπόλοιποι συνάδελφοι πιστεύουν ότι η προστασία των πελατών είναι σημαντικό θέμα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και πιστεύω ότι φαίνεται ότι υπάρχει ένα κοινό θέμα για μεγαλύτερη διαφάνεια και αναλογικότητα. Και φυσικά μπορώ να το υποστηρίξω αυτά. Υπάρχουν ε, και αναφορές ε, στις τροπολογίες, ε, στις εργασίες που πρέπει να γίνουν σε διεθνές επίπεδο, κάτι που μας βοηθά να λάβουμε υπόψη στο συστημική, συστημική φύση των κεντρικών αντισυμβαλωμένων. Σε ό,τι αφορά τα διάφορα μεγέθη και τη φύση των κεντρικών αντισυμβαλωμένων, υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των μεγάλων και των μικρών αντισυμβαλωμένων. Κάποιες από αυτές τις τροπολογίες προσπαθούν να αναγνωρίσουν τις διαφορές μεταξύ τους. Σε άλλου τομεί, όπως αναμένεται, υπάρχουν και άλλοι τομείς αποκλήσεων. Δεν θέλω να καθυστερήσω ε, πάρα πολύ γιατί εφού υπάρχουν διάφορες αποκλήσεις ε, μπορεί να σημαίνει ότι κάποια συγκεκριμένη γραμμή ακολουθείται από κάποιο βουλευτή ή ομάδες. Θα ήθελα να ακούσω βέβαια τους συναδέλφους, ε, ίσως να μπορέσουν να με πείσουν. Υπάρχουν πολλές ε, τροπολογίες ε, που προσπαθούν να κάνουν μια σαφή διάκριση ε, μεταξύ των σεναρίων αθέτησης και μη αθέτησης υποχρέωσης και όλα καταλήγουν στα ίδια συμπεράσματα, αλλά θέλουν μεγαλύτερη σαφήνεια μεταξύ αυτών των δύο τρόπων με τον, στους οποίους μπορεί κάποιος να μπλέξει ως κεντρικός αντισυμβαλωνόμενος. Είναι λοιπόν καλό με τους σκιώδεις τώρα να συνεργαστούμε για να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά και πού μπορούμε να καταλήψουμε. Γιατί Όλοι συμφωνούμε ότι αν έχουμε διαφάνεια και σαφήνεια θα βοηθήσει αυτό το σύστημα. Στην 2.31 ε, προσπάθησα να αναφερθώ στην ε, ε, σαφή ελληλουχία της χρήσης των εργαλείων της διάσωση, θα πρέπει να περιορίσουμε ε, το hair cutting και ε, ένα τελευταίο εργαλείο ε, είναι ουσιαστικά κάτι που θα πρέπει να δούμε όταν υπάρχει μια γκρίζα ζώνη μεταξύ εξυγίανσης και ανάκαμψης και στη 2.37 προσπάθησα να δώσω σαφήνεια ότι στο αρχικό περιθώριο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καθαριστικά μέλη που δεν ευθύνουν τις υποχρεώσεις υποχρεώσεις δηλαδή να είμαστε σίγουροι ότι ε, τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών δεν θα χρησιμοποιηθούν εκτός ε, και αν μπούμε σε διαδικασία εξυγίανσης και κατόπιν η αρχή της εξυγίανσης θα κάνει αυτά που πρέπει. Χαίρομαι που είδα ότι κάποιοι συνάδελφοι από τους φιλελευθέρους και τους πρεσίνουν ε, περιορίζουν την χρήση του UMGIH περαιτέρω περιορισμοί για ε, το πότε ε, θα χρησιμοποιούμε το αρχικό περιθώριο και το haircutting, το κούρεμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, εγώ έχω τονίσει κάποιες διαφορές. Επίσης, το stress test ήρθε κάποια στιγμή αργότερα, κατόπιν των τροπολογιών. Προσπάθησα εγώ να βάλω την τροπολογία δεν 99 που καλεί ε, να έχουμε τακτικά stress test ε, και τέτοια εγχειρήματα να υλοποιούνται και υπάρχει ρόλος και για την Εθνική Αρχή που είναι ο σημερινός επόπτης ε, και φυσικά και τα σώματα εξυγίανσης ε, μπορούν να συμμετέχουν ε, σε ε, συνεργασία με την EACB. Και μάλιστα θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι γνωρίζουν ποια θα είναι τα αποτελέσματα στην οικονομική σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ρόλους για τις εθνικές αρχές θα συζητήσω με τους συναδέλφους για αυτό το θέμα. Για το NCWO είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα και στην ε, τροπολογία μου 436 ε, προσπαθώ να ορίσω το NCWO ε, και πώς αυτό θα στεκόταν σε ένα δικαστήριο. Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στην αρχή εξυγίανσης να δράσει εφαρμόζοντας μια σαφή αρχή NCWO για να μπορεί να δράσει χωρίς επιφυλάξεις αν αντιμετωπίσει ε, νομικά προβλήματα θα είναι καλό να υπάρχει αυτή η διάταξη. Υπάρχει ένα σύνολο στοιχείων που έχουν υποβάλει οι συνάδελφοι. Θέλω να τα δούμε και να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε το NCWO και να δούμε τι ακριβώ θα κάνουμε μέσω αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν και άλλε αποκλίνουσε απόψει σε σχέση με τον συμψηφισμό. Ε, εδώ ε, οι κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι πελάτες ε, λαμβάνουν την κατάλληλη αποζημίωση αν χρησιμοποιηθούν τα περισσοκά του στοιχεία για τη διαδικασία της εξυγίανσης, της ανάκαμψης. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στα οποία συμφωνούμε, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά σημεία επί των οποίων μπορούμε να συνεργαστούμε και ανυπομονώ να συνεργαστούμε και με τον συγγητή, όπως κάνουμε και τους τελευταίους μήνες, αλλά να προσπαθήσουμε και με τους σκιώδεις να βρούμε συνένεση σε ένα τεχνικό φάκελο, αλλά πάρα πολύ σημαντικό. Και ελπίζω ότι ακόμη και αν νομοθετήσουμε δεν θα χρειαστεί ποτέ να τεθεί σε εφαρμογή. Ευχαριστώ, Κέι. Να δώσω το λόγο τώρα στον ε, συνεισηγητή, στον Γιάκομπ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι συνολικά όταν εξετάσαμε τις τροπολογίες συνειδητοποιήσαμε ότι η Κέι και εγώ θα έχουμε ένα σχετικά εύκολο έργο μπροστά μας. Πρώτον, γιατί πολλές από τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί αποτελούν ενδιαφέρουσες προσθήκες σε αυτό που έχουμε εμείς προετοιμάσει στην έκθεσή μας. Για παράδειγμα, υπήρχαν κάποιες προσθήκες από τους πράσινους όσον αφορά μια διαρκή δοκιμή ε, σε σενάρια ακραίων καταστάσεων, Τροπολογία από το ΕΛΚ για το τι θα γίνει σε περίπτωση παράβασης των κανόνων και στην, στην έκθεση μας πράγματι δεν λαμβάναμε υπόψη μας ε, ε επαρκώς αυτό το θέμα. Υπάρχουν σχετικές διατάξεις στον κανονισμό BRRD, αλλά μπορούμε να, το, να, να εντάξουμε τέτοιες διατάξεις και εδώ. Είπε και η ΚΕΙ και περιέγραψε τους ε, τομείς όπου υπάρχει σύγκληση ε, απόψεων. Δεν θα επαναλάβω εκείνα που εκείνη είπε. Θέλω όμως να κάνω κάποια σχόλια για τρεις τομείς όπου υπάρχει διαφωνία. Ε, πρώτον, όσον αφορά την ίση μεταχείριση των πιστωτών. Εδώ πρέπει να συμπεριληφθούν τα συστημικά αποτελέσματα. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι θα ακολουθείται σε μια χώρα αυτή μια διαδικασία εξιγής ε, καθάρισης ε, σε μια συγκεκριμένη χώρα ενώ στον υπόλοιπο κόσμο δεν θα συμβαίνει τίποτα, θα είναι σαν να μην έχει ε, προηγηθεί το οτιδήποτε. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί λοιπόν γιατί αν δεν είμαστε προσεκτικοί θα καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου παρά την, ε, συμφωνία όλων ότι ε, οι φορολογούμενοι θα είναι η έσχατη λύση θα καλούνται οι φορολογούμενοι τελικά να αποζημιώνουν ε, ιδιώτες ε, αυτό είναι κάτι που προφανώς δεν θα έπαιρνε υπόψη αυτόν τον συστημικό χαρακτήρα. Δεύτερον, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για την αποζημίωση. Στην έκθεσή μας η ΚΕΙ και εγώ καταθέσαμε πρόταση για την αποζημίωση σε περίπτωση ανάκαμψης, στο πλαίσιο της ανάκαμψης, με σκοπό όλοι οι ιδιώτες που εμπλέκονται, τα καθαριστικά μέλη, κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι και οι πελάτες έχουν κοινό συμφέρον από την επιτυχή κατάληξη της ανάκαμψης και από την διάσωση, την επιβίωση του κεντρικού αντισυμβαλωμένου. Αυτό πρέπει να διατηρηθεί. Ταυτόχρονα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι από τη στιγμή που ε, ξεπεράσεις την, την, την ανάκαμψη και περάσεις σε εξυγίανση υπάρχουν δύο βασικοί στόχοι όπου οι κρατικές ή ευρωπαϊκές αρχές πρέπει να, ε, να εξυπηρετήσουν πρώτον να διασφαλίσουν τα συμφέροντα των φορολογουμένων και να εξασφαλίσουν τη συστημική σταθερότητα ε, της οικονομίας και ε, τα καθαριστικά μέλη και οι πελάτες θα πρέπει να αποφύγουν καταστάσεις όπου ε, τα δικά του συμφέροντα δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά την ε, εξυγίανση. Γι' αυτό και στην, ε, στη φάση της εξυγίανσης θα, θα, πρέπει να μην αποζημιώνονται οι, οι τρεις αυτοί εμπλεκόμενοι. Και τελευταίο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι έχουμε μια ε, τεράστια ευκαιρία, όχι μόνο ως προς την ανάκαμψη, γενικότερα να κινηθούμε προς μια ενιαία αρχιτεκτονική εποπτείας. Η μεγάλη κεντρική αντισυμβαλόμενη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η η, οι κατεξοχήν συστημικοί παίκτες στην χρηματοπιστωτική αγορά και θα υπάρξουν ε, σοβαρά διασυνοριακά προβλήματα αν συνεχίσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζήματα σε εθνικό επίπεδο. Είναι πολύ ευκολότερο να δημιουργηθεί μια ενιαία αρχή σε αυτόν τον τομέα από ό,τι ε, ήταν για την ε, ενιαία τραπεζική αρχή, διότι ο αριθμός των κεντρικών αντισυμβαλλωμένων είναι πολύ μικρός, είναι πέντε ίσως και λιγότεροι. Άρα δεν θα είναι δύσκολο να αξιοποιήσουμε αυτό το στοιχείο και να καταλήξουμε ε, σε κατάσταση ε, όπου δεν θα μπορεί ε, η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Μάλτας να βρίσκεται υπό ευρωπαϊκή εποπτεία ενώ άλλοι κεντρικοί της συμβαλόμενοι με δεκάδες τρισεκατομμύρια χαρτοφυλάκια να διαχειρίζονται να μην υπόκεινται σε καμία εποπτεία. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Όχι μόνο η εποπτεία λοιπόν πρέπει να μας απασχολήσει, αλλά και η ενιαία διαδικασία ανάκαμψης και εξυγίανσης. Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Έκανα λοιπόν ε, μια πρόταση στις τροπολογίες μου σχετικά με την ανάγκη να υπάρχει ένα κεντρικό ενιαίο ταμείο ανάκαμψης. Αυτά βεβαίως είναι θέματα που υπερβαίνουν το, το, αυτού του συγκεκριμένου θέματος είναι, ε, ε, έχουν ένα ευρύτερο χαρακτήρα αυτά τα θέματα. Ε, εν πάση περιπτώσει θα ήθελα παρόλα αυτά να ευχαριστήσω την συνεισηγήτρια και τους ε, Ευχαριστώ. Ξεκινήσουμε με την κυρία Ντανούτα Χιούμπνερ, σκιώδη του ΕΛΚ. Ευχαριστώ Μάρκους. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι από την αρχή στη διάρκεια των συζητήσεων που είχαμε αλλά και σε αυτό το τελικό επιτέλεσμα, την έκθεση, ε, συμμερίζομαι την ε, προσέγγιση των συνεισηγητών και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω και για το γεγονός ότι έλαβαν υπόψη τους αυτά που λέγαμε ε, στις συναντήσεις μας πριν από την οριστικοποίηση του κειμένου τους. Ξέρω ότι η πρόταση της Κομισιόν ήταν γενικά καλή. Παρ' αυτά ήταν δύσκολο το θέμα αυτό, τεχνικό ε, όμως ε, έφερνε, άφηνε ανοιχτά πολλά ενδεχόμενα, πολλές επιλογές και έτσι η δουλειά της Κέι και του Γιάκοπ ε, ήταν εξαιρετική. Ελπίζω να συνεχιστούν αυτές οι θετικές συζητήσεις ε, κατά τη διαδικασία επεξεργασίας των συμβαστικών τροπολογιών. Να σας παρουσιάσω λίγο τις τροπολογίες που κατέθεσα εγώ. Κάποιες από αυτές επικεντρώνονται στην προβλεψιμότητα, την σαφήνεια, την νομική βεβαιότητα, την ασφάλεια δικαίου, ιδίως όσον αφορά τα σχέδια ανάκαμψης. Και εδώ προτείνω να υπάρχουν κάποιες έντολες για τον ΕΣΜΑ, ε, για την κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων ε, ή την ε, ε, Στου τομεί όπου ήδη προβλέπεται από τον κανονισμό BRRD, αλλά δεν προβλέπονται στην πρόταση αυτού του κανονισμού. Επίσης, προτείνω ε, οδηγίες και τευτήριε γραμμέ να προέρχονται από τις διεθνείς εργασίες όσον αφορά τα σχέδια ανάκαμψης και τα σενάρια που θα προβλέπονται, καθώς και τις κατηγορίες εργαλείων που θα κατοχυρώνονται και, τέλος όσον αφορά την σαφήνεια ε, προτείνω κάποιες ε, προσθήκες ε, για να αποσαφινιστεί να αποσαφινιστεί διάκριση μεταξύ περιπτώσεων αθέτησης και μη αθέτησης. Όσον αφορά την ενίσχυση ε, των διατάξεων για το δημόσιο χρήμα υπέβαλα κάποιες τροπολογίες για να ξεκαθαριστεί ότι τα χρήματα των φορολογουμένων πραγματικά θα είναι η έσχατη λύση. Επίσης, για την, ε, για την αναστολή των ε, υποχρεώσεων εκαθάρισης. Προτείνω ότι θα πρέπει αυτή να ε, εφαρμόζεται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και από τεχνικής άποψης προτείνω και κάποιες τροπολογίες για διοικητικά πρόστιμα που βεβαίως προβλέπονται και από την πρόταση της Κομισιόν αλλά μέσω τροπολογιών στην, ε, στον κανονισμό BRD ε, και νομίζω ότι θα πρέπει να ενταχθούν και εδώ. Θα συνεχιστούν βεβαίως οι συζητήσεις για τα ζητήματα στα οποία δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει συμφωνία. Η πρόθεσή μου γενικά είναι να καταλήξουμε σε ένα σύστημα δεδομένου ε, του, της διαδικασίας ε, αναθεώρησης του πλαισίου λειτουργίας των κεντρικών συμβαλωμένων θα είναι προσωρινό έως ότου καταλήξουμε σε ένα πιο μόνιμο ε, καθεστώς. Ε, προτείνω για παράδειγμα να συμμετέχουν ε, στα κολέγια εξυγίανσης εκπρόσωποι των μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ε, ως παρατηρητές. Βεβαίως αυτό επιβαρύνει την όλη διαδικασία, την καθιστά πιο δύσκολη, αλλά παρόλα αυτά εξασφαλίζει ότι ε, ε, δεν θα υπάρξουν ε, καταχρήσεις ή καθυστερήσεις. Επίσης, προτείνω και κάποια στοιχεία που υπάρχουν και στο πλαίσιο ΕΜΙΡ. Ξέρω ότι η δομή του, του, του κολεγίου είναι ε, ε, δύσκολη και βαριά, ε, γι' αυτό και προτείνω μια ρήτρα αναθεώρησης για ε, το συνολικό σύστημα ε, των διαδικασιών εξυγίανσης να μπορούν δηλαδή να αναθεωρούνται οι ισχύουσες, οι ισχύοντες κανόνες αν κρίνεται αναγκαίο. Επίσης, συμφωνώ με την πρόταση των εισηγητών να προβλέπεται ένα κεφάλαιο κεντρικού αντισυμβαλωμένου ως πρώτη λύση, ως πρωτού ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία ανάκαμψης εξηγήσεις και ε, προτείνω συγκεκριμένα να βαθμονομείται αυτό το κεφάλαιο με τον, ε, με τον πλέον ισορροπημένο ε, τρόπο. Και να πω και κάτι τελευταίο. Επειδή γνωρίζω ότι θα είναι δύσκολο Θέλω όμως να υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής το, των, της ε, συμμετοχής των κεντρικών αντισυμβαλωμένων, να υπάρχει δυνατότητα ε, συζήτησης ε, και των, όσον αφορά τα αμοιβαία κεφάλαια που ναι, θα συνεισφέρουν οι κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι. Και καθώς βρισκόμαστε στο μέσο της διαδικασίας συζητήσεων και διαβουλεύσεων, προτείνω να υπάρχει δικαίωμα αποζημίωσης των, ε, ε, ε, των πελατών και των μελών εκαθάρισης στην εξυγίανση και, αλλά όχι στην ανάκαμψη προκειμένου να αναγνωρίζεται η, η, σημασία που έχει να στέφεται με επιτυχία η ανάκαμψη. Θα συνεχιστούν οι συζητήσεις. Η μεταχείριση πιστωτών. Εγώ αναδιοτύπωσα αυτό που νομίζω ότι ήταν πρόθεση της Κομισιόν και που βεβαίως ευθυγραμμίζεται και με το έργο του SFB. Προτείνω να μην περιλαμβάνονται τα, να μην περιλαμβάνεται το κόστος αν, αντικατάστασης. Έχουν γίνει καλές συζητήσεις ε, έως, αυτό το, ως προς αυτό το θέμα είναι γεγονός ότι ε, μια ισχυρή βάση μπορεί να ε, ε, δημιουργηθεί μόνο όταν τα επιμέρους στοιχεία μπορούν να μετρούνται με συγκεκριμένο τρόπο, με ακρίβεια και όσον αφορά την η αβεβαιότητα, πρέπει να αρθεί αυτή η αβεβαιότητα όσον αφορά το, τις δαπάνες αντικατάστασης και ακριβώς αυτό το, το στόχο εξυπηρετούν οι τροπολογίες μου. Βεβαίω, όπω είπα, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν και είμαι βέβαιη ε, ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή λύση, καθώς φαίνεται ότι υπάρχει διαφωνία. Ε, όχι μόνο εδώ μέσα, αλλά και μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, των ε, φορέων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Ευχαριστώ, φιλελεύθερη. Παρακαλώ. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο ε, ξεκίνησα ως Ευρωβουλευτής, οπότε είμαι πολύ καινούρια. Οπότε δεν μπόρεσα να συμμετάσχω στη συζήτηση στη δεύτερη εβδομάδα για αυτούς τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους και την ανάκαμψη και εξυγίανση. Ε, οπότε ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους και ιδιαίτερα του προκατόχου μου και θα διαμορφώσω άποψη τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο που κατέθεσε τις τροπολογίες μας και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για το θέμα αυτό. Εμείς ως Άλντε θέλουμε να ενισχύσουμε το κείμενο μέσω των τροπολογιών μας για τη χρήση λοιπόν δημοσίων πόρων η συνδεσιμότητα των CCP, των κεντρικών αντισυμβαλωμένων και η σωστή λειτουργία του ότι κανείς πιστωτής δεν θα πρέπει να υποστεί μία. Το NCWO είναι, είναι βασικό για να μην χρειαστεί να εισρεύσουν ε, δημόσιοι πόροι, οι οποίοι θα πρέπει μόνο να εισρεύσουν αν είναι απόλυτα αναγκαίο για να αποφευθεί μια ε, γενικευμένη συστημική κρίση και θα θέλαμε να είναι δυνατόν να ε, επιστραφούν ε, οι δημόσιοι πόροι που θα έχουν χορηγηθεί από τους ε, πιο εύπορους από τα πιο εύπορα αντισυμβαλόμενα μέρη. Επίσης, επειδή αυτά τα CCP είναι άλλο συνδεδεμένα, μπορεί ένα πρόβλημα σε ένα CCP να επηρεάσει και τα άλλα. Πρέπει λοιπόν να αναλύσουμε σωστά την ε, σύνδεση των CCP με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και γενικότερα ε, τι ρόλο παίζουν στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα. Και γι' αυτό υποβάλαμε τροπολογίες, ούτω ώστε αν υπάρχει κύβερνο απειλή να συμπεριληφθεί και αυτή. Επιπλέον, οι τροπολογίες μας προβλέπουν ε, ένα ευρύτερο ρόλο και για την ΕΜΣΑ, για παράδειγμα, για την κατάρτιση των σχεδίων ανάκαμψης. Επίσης, η αρχή NCWO είναι βασική για να είναι ισορροπημένη η νομοθεσία και το οποιοδήποτε σχέδιο ανάκαμψης πρέπει να το λάβει υπόψη του. Όλα αυτά πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένα ώστε η αρχή εξηγένσης να έχει χώρο ελιγμών. Υποβάλλουμε λοιπόν μια τροπολογία για να υπάρχει δυνατότητα επιστροφής των δημοσίων πόρων και ε, αυτά, αυτοί οι πόροι να χρησιμοποιηθούν για την χρήση, για την, συγγνώμη, για την αποζημίωση των ε, πιστωτών που θα έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη ζημία. Για την τροπολογία για τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης τώρα δεν νομίζω ότι έχει έννοια να το συζητήσουμε αυτό όταν θα συζητήσουμε το ΕΜΙΡ. Πολλά έχουμε ακόμη να συζητήσουμε ως ε, σκιώδης και φυσικά προσβλέπω να συμμετάσχω στην ευρία πλειοψηφία που πρέπει να διαμορφωθεί για αυτό το σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ πολύ για την ΚΟΕ. Δεν είναι εδώ ο Μιγέλ. Αλλά ποιος τον αντικαθιστά. Ευχαριστώ να πω κάτι αντί για το Βιέγκα. Μου είπε να εκπροσωπήσω σήμερα την ομάδα μας αλλά πρέπει καταρχάς να τον ευχαριστήσω για την ε, συνεργασία για το θέμα αυτό, το τόσο σημαντικό. Εδώ έχουμε, είναι γνωστό, διαφορετικές απόψεις. Συμφωνούμε ότι δεν θα πρέπει να πληρώνουν οι φορολογούμενοι τις αποτυχίες των αγορών. Αυτό άκουσα και από την ε, εισαγωγή της ε, εισηγήτριας και όπως ξέρετε ο κύριος Βιέγκα θα συμμετάσχει ε, κατόπιν ε, όταν θα επανέλθει. Να σας διαβάσω τώρα τους, ε, τις παρατηρήσεις του. Στοχεύουμε με τις τροπολογίες μας να μην πληρώσουν οι φορολογούμενοι τις, απολυ... τις αποτυχίες διαφόρων ιδιωτικών φορέων, είτε είναι CCP είτε κεντρική αντισυμβαλόμενη. Πρέπει λοιπόν η αρμόδια αρχή ανάκαψης να μπορεί να παρεύει εγκαίρως. Δεν θα πρέπει να περιοριστούν οι εξουσίες της. Εάν υπάρξουν δημόσιοι πόροι για να διασωθεί ένα CCP, είναι λογικό ότι θα πρέπει να μεταφερθούν στο κοινό ε, όλες οι σχέσεις ιδιοκτησίας, χωρίς ε, κανένα περιορισμό και όρο. Δεν συμφωνούμε ότι η δημόσια ε, ιδιοκτησία κάποιων τέτοιων οργανισμών θα πρέπει να είναι προσωρινή θεωρούμε ότι έχουμε ήδη συμβατικούς, ε, συμβατικές δυνατότητες για την ανάκαμψη και εξυγένση και θα πρέπει να υπάρχουν και περισσότερες δυνατότητες για νωρίτερη παρέμβαση. Η αρχή εξυγένσης θα πρέπει να απαιτεί ε, ισχυρές κεφαλιακές απαιτήσει από τα CCP πέρα και από το ΕΜΗΡ και να ζητάει και αλλαγές στην ιδιοκτησιακή δομή το CCP αν χρειάζεται. Δεν νομίζουμε ότι τα CCP, επειδή διαχειρίζονται κινδύνους, είναι, θα πρέπει να είναι υπεύθυνα για τους κινδύνους των ε, μελών ή οποιονδήποτε ιδιωτικών πελατών όταν κάνουν συναλλαγές. Θα πρέπει οι πελάτες να είναι υπεύθυνοι για τους κινδύνους που αναλαμβάνουν. Θα πρέπει να υπάρχουν επαρκείς μηχανισμοί για την κατανομή αυτών των κινδύνων και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στους πρασίνους. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους δύο εισηγητές. Είναι πολύ καλό παράδειγμα να λειτουργεί καλά η ευρωπαϊκή χαράξη πολιτικής και έχουμε τις καλύτερες προτάσεις από όλες τις ομάδες. Ίσως ε, ε, η ΚΕΙ μάλλον θα συμφωνεί μαζί μου ότι δεν θα συνεχίσουμε να ασκούμε έτσι πολιτική. Θέλω να καλωσορίσω και την Καρολάιν. Καλώς ήρθατε, αν και μπαίνετε σε βαθιά νερά. Εμεί από την πλευρά του Πρασίνων καλωσορίζουμε την πρόταση και πιστεύουμε ότι έχει λογική το σχέδιο έκθεση. Όμω ε, θα εξετάσουμε φυσικά τι τροπολογίε που έχουν προταθεί. Θα μιλήσω για τι ε, τροπολογίε που προωθούμε εμεί. Ε, στην 263 για την αιτιολογική σκέψη 60. Θεωρούμε ότι οι κυβερνήσει θα πρέπει κάποιε φορέ να παρεμβαίνουν όταν πιστεύουν ότι δεν λειτουργεί η εξυγίανση, αλλά δεν πιστεύουμε, όπως και στην BRRD, ότι θα πρέπει να λέμε πώ θα το κάνουμε κάνουμε αυτό, καθώς μιλάμε για το πλαίσιο ανάκαμψης και εξυγίανσης, ε, έχει σχεδιαστεί για να μην εμπλέκονται οι φορολογούμενοι θα δεχόμαστε μία διάταξη ότι ε, θα πρέπει να αιτιολογείται η χρήση εργαλείων μη εξυγίανσης, ε, όμως ε, πολύ συχνά το να αναλαμβάνει κάποιος τις δικές, να μην αναλαμβάνει τις φορολογικές του ευθύνες σημαίνει ότι παρεμβαίνει σε δημοσιονομικές ευθύνες άλλων κρατών μελών. Τώρα, γιατί να μην διατηρήσουμε του ρόλους και τις ευθύνες όσο δυνατόν πιο σαφείς απαιτώντα μία αρχή να παρεμβαίνει Πιστεύουμε ότι η ανεξαρτησία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων ε, είναι πολύ πιο αδύναμη από ότι η επιχειρησιακή ανεξαρτησία, οι συγκρούσει ε, συμφερόντων ε, ουσιαστικά θα έρθουν και θα παρέμβουν εδώ. Στην 369 δηλώνουμε ότι θα πρέπει το σχέδιο εξυγίανσης να συνάδει με τα σχέδια των κρατών μελών και ε, των εκαθαριστικών μελών. Ε, σε περίπτωση σενερίου μπορεί να υπάρχει παράλληλη εξυγίανση του CCP και ενό εκαθαριστικού μέλου τουλάχιστον. Πρωτεύουμε νέα διατύπωση στην 459 να έχουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα οι CCP να εφαρμόσουν τα μέτρα σύμφωνα με τι απαιτήσει που έχουμε στα άρθρο είναι απαραίτητο να θέσουμε ένα ε, όριο, μια προθεσμία για το στάδιο της προεξυγίανσης και αν δεν δούμε παρκή αποτελέσματα τότε θα πρέπει να ξεκινήσει η εξυγίανση. Η τροπολογία μας 560 υποστηρίζει την 561 του Γιάκοπ, αλλά προσθέτει και άλλη προστασία έναντι πιθανών απαιτήσεων που θα είχαν οι πιστωτές ε, ή θα είχαν υφεστεί απώλειες επειδή ε, μπορεί να είχε μεταφερθεί ένα μέρος ε, των επιχειρήσεων σε μια βιώσιμη οντότητα. Τώρα σε για όσους εκτίθεται πιστεύουμε ότι πρέπει ο κεντρικός της τουλάχιστον καθημερινά να ε, κάνει μια αξιολόγηση για πιθανές απώλειες για τους λόγους ε, του περιθωρίου. Ε, πρέπει να ε, χρησιμοποιούνται οι κατάλληλοι αλγόριθμοι ε, σε πολύ συχνή βάση, όμως αυτό αντισταθμίζεται ε, αν διαχειρίζονται οι χρήστες του ECP κατα, καταλήλως τους κινδύνους. Επιστηρίζουμε την ιδέα να είναι επικεφαλής η ΕΣΜΑ για τα stress test, αν δούμε την ευρύτερη εικόνα. Πιστεύω λοιπόν ότι γενικά συμφωνούμε, όμως υπάρχουν και πολλές ευκαιρίες για να συζητήσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στις συναντήσεις των σκιωδών και ανυπομονώ. Ευχαριστώ μόλι. Δεν βλέπω τον, τον κύριο Μονό, δεν είναι εδώ. Φτάνουμε στο Κατσιγιάι λοιπόν. Βλέπω ποιος δεν έχει μιλήσει ακόμη. Παρακαλώ, κύριε Μπερές. Ευχαριστώ. Πολλά υπόθηκαν από τους ε, εισηγητές και τους κοιόδης. Δεν θα με ίσως να εξηγήσω εγώ στη βάση ποιου πνεύματος έχω καταθέσει κάποιες ε, τροπολογίες ή έχω συνυπογράψει κάποιες τροπολογίες. Υπάρχει ε, μια σειρά τροπολογιών που καλύπτουν κάποιες ανησυχίες της Κεντρικής Τράπεζας σε ένα βαθμό συμφωνούμε με τους συνεισηγητές, αλλά σε κάποια άλλα σημεία νομίζω ότι είναι καλό να διαχωρίσουμε και να αποσαφηνίσουμε τις ευθύνες της κάθε αρχής και να ξεκαθαρίσουμε τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών και της ίδιας της Κεντρικής Τράπεζας. Υπάρχει και ένα σημείο στο οποίο θέλω να επανέλθω πιο συγκεκριμένα. Αυτό έχει να κάνει με το πνεύμα των τροπολογιών μου. Το πρώτο έχει να κάνει με τους τελικούς πελάτες. Γιατί στην ε, εξυγίανση λαμβάνονται πλήρω υπόψη τα συμφέροντα των τελικών πελετών, όμως μπορεί να υπάρχει ο κίνδυνος να εμποδίσουμε την ίδια τη διαδικασία της εξυγίανσης. Έτσι λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε το εξής. Γενικά, ε, αναφερόμαστε και επικαλούμαστε μία αποζημίωση και αναφερόμαστε στους τελικούς πελάτες, εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Όμως τη στιγμή που η ίδια η εξυγίανση θα πρέπει να γίνει υποπλήρη διαφάνεια και με κατάλληλο χειρισμό των τελικών πελατών μπορεί τελικά να εμποδίσουμε την ίδια τη διαδικασία της εξυγίανσης να λάβει χώρα. Ακόμη και την ανάκαμψη. όπως είπαν και άλλοι ομιλητές, και εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε λίγο παραπάνω τις προτάσεις έτσι ώστε να δίνονται κίνητρα σε κάποιους να πάνε προς την ανάκαμψη και την εξυγίανση. Και ο σκοπός εδώ είναι να αποφευχθεί η χρεοκοπία, η αθέτηση της υποχρέωσης και φυσικά να γίνει με αυτή τη σειρά πρώτα να έχουμε την ανάκαμψη και μετά την εξυγίανση. Υπάρχουν ε, και κάποιες τροπολογίες που κατέθεσα και σκοπεύουν στο να δώσουν ε, μεγαλύτερη ευελιξία στις ε, αρχές εξυγίανσης. Εδώ τετραγωνίζουμε τον κύκλο τέλος πάντων, γιατί αφενός θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι αρχές εξυγίανσης δεν θα κάνουν αυθαιρεσίες, αλλά απ' την άλλη θέλουμε να μπορούν να προσαρμοστούν στις συνθήκες που έχουν να αντιμετωπίσουν και να διαθέτουν μια πλήρη εργαλειοθήκη χωρίς να υπάρχουν και πάρα πολλοί περιορισμοί. Δηλαδή χωρίς να είναι όλα προκαθορισμένα. Ένα τελευταίο σημείο έχει να κάνει με τις τρίτες χώρες. Εδώ πιστεύω ότι πήγαν κάπως μακριά οι δύο εισηγητές και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχουμε τους κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη σκοπιά αυτή ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη και μία συζήτηση στο διεθνές επίπεδο για τα διεθνή πρότυπα. Θα πρέπει να ενταχθεί και αυτό στους προβληματισμούς μας, γιατί και η Κεντρική Τράπεζα έχει τέτοιες ανησυχίες που τις θεωρώ νόμιμες. Υπάρχει και μια συζήτηση που αναφερθήκε μια συζητηση που και απο την συνάδελφο από τους Φιλελευθέριους για αν θα πρέπει να έχουμε μια ενιαία ε, αρχή εξυγίανσης, ε, ένα νέο και τα κτλ. Συνεχίζονται αυτές οι συζητήσεις σε διεθνές επίπεδο και όταν εμείς ως Επιτροπή συναντήσαμε τις αρχές του Συμβουλίου Χρηματοπιστήτης Σταθερότητας του FSB στη Βασιλεία, κάναμε μια ανταλλαγή απόψεων ε, και νομίζω ότι μα νομιμοποιεί να έχουμε μια ρήτρα αναθεώρησης πιο λεπτομερή ως ε, προς ε, την ε, ένταξη της δυναμικής αυτής της συζήτησης στις θέσεις που αποτυπώνονται. Και κάτι τελευταίο. Επαναλαμβάνω κάτι που έχω πει σε περασμένη συνεδρίαση. Νομίζω ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε μια αρκετά ρεαλιστική προσέγγιση και πιστεύω ότι η προσέγγιση των δύο συνεισηγητών, αυτή που μας προτείνει στο αρχικό κείμενο, για να μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο και χωρίς χρονοτριβή να έχουμε ένα σύστημα ανάκαμψης και εξυγίανσης των κεντρικών αντισυμβαλωμένων, ε, χωρίς να το συνδέσουμε με όλους τους άλλους φακέλους που έχουμε επιτάπητος. Γιατί διαφορετικά θα έχουμε συστήματα τα οποία θα αυτομπλοκάρονται ενώ υπάρχει πραγματική ανάγκη να υπάρξουν τα συστήματα αυτά. Κοιτάξτε, αν υπάρχει αυτό το σύστημα εξυγίανσης ε, ε, και ανάκαμψης, να το σκεφτούμε, γιατί χρειαζόμαστε αυτή την ομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ. Σάντερ, παρακαλώ. Merci, euh, Monsieur le Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους ε, εισηγητές. Πολλά υπόθηκαν. Θα πάρω κι εγώ εν συντομία το λόγο για να τονίσω δύο σημεία. Το πρώτο έχει να κάνει με την αναγκαιότητα και οι κανόνες διαχείρισης και εξυγίανσης ε, να είναι αρκετά ευέλικτοι. Αυτό έτσι ώστε οι αρχές εξυγένσης να μπορούν να λάβουν τις καλύτερες αποφάσεις σε ένα χρηματοοικονομικό περιβάλλον που μπορεί να είναι ασταθές. Το δεύτερο σημείο που θέλω να τονίσω έχει να κάνει με την αναγκαιότητα να δούμε πολύ προσεκτικά τις πτυχές τρίτη χώρα, τρίτες χώρες. Αυτά είναι τα δύο σημεία επί των οποίων ήθελα να επιμείνω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καθώς έχουμε χρόνο, θα ήθελα να δώσουμε το λόγο στον Πάτρικ Πίρσον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα θα μιλήσω. Να σας καλωσορίσω σε αυτό το μαγικό κόσμο των ε, CCP, CM και ιδιωτών πελατών. Τεχνικές ε, τροπολογίες. Τις χαιρετίζουμε και είμαστε απολύτως ανοιχτοί σε βελτιώσεις και βλέπουμε ότι ο διάλογος μεταξύ των ευρωβουλευτών και του κλάδου της οικονομίας και άλλων εμπειρογνωμένων έχει οδηγήσει σε πολλές τροπολογίες για τη βελτίωση και την αποσαφήνιση της αρχής πρότασης της Κομισιόν και το χαιρετίζουμε αυτό. Επίσης, ε, δεν θέλουμε να αποκλίνουμε πολύ από τις ζητήσεις που γίνονται στο Συμβούλιο μεταξύ των κρατών μελών. Θέλω να θέσω πέντε σημεία όπου πιστεύω ότι πρέπει να γίνει περαιτέρω συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη και τις συζητήσεις που γίνονται στο Συμβούλιο επί της πρότασης Κομισιόν. Το πρώτο αφορά το, το, το ότι θα πρέπει πρώτα να επιβαρύνονται οι CCP ως προς τις ζημίες. Υποστηρίζουμε ως Κομισιόν τρία ζητήματα. Υπάρχει, ε, χρειάζεται, χρειαζόμαστε μια, ένα δεύτερο επίπεδο ε, απορρόφησης ζημιών. Ε, έχει προταθεί αυτό. Εμείς έχουμε κάποιες αμφιβολίες, διότι αυτό αφορά και το κεφάλαιο που παραμένει στους κεντρικούς ανζυμβολημένου και το οποίο θα εξαντληθεί πλήρως σε περίπτωση αθέτησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έχει, είναι, είναι μόνη δικαιοδοσία στον κόσμο όπου υπάρχει μία και μόνη ένα, ένα στρώμα απορρόφησης ζημιών το να, το να εισαχθεί και ένα δεύτερο, μια δεύτερη γραμμή ε, άμυνας ε, είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα αλλά δεν πρέπει να αποκλίνουμε πολύ από το τι συμβαίνει ε, ε, στον υπόλοιπο κόσμο. για τις δομές των ομίλων. Ε, τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση που έχουν κεντρικό αντισυμβαλόμενο. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχουν επιπτώσεις λόγω διαφορετικών εταιρικών δομών στα διάφορα κράτη-μέλη και πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς ε, ως προς το ποια είναι η πρόθεσή μας. Ενδεχομένως δεν υπάρχει πανάκια. Δεν υπάρχει κάποια, κάποια διάταξη που θα μπορούσε να λειτουργήσει ω πανάκια σε όλες τις περιπτώσεις δηλαδή. Επιβάρυνση κατά, κατά κύριο λόγο του ε, CCP. Μιλάμε για, την, για τα σχέδια ανάκαμψης. Ε, δεν ξέρω αν είναι ε, ε καινοτομία ε, ε, πάντως είναι σε κάθε περίπτωση κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναεξετάσει και θέλουμε περισσότερο χρόνο για να, το συζητήσουμε πώς θα, μπορούσε αυτή η, η καινοτομία ε, να ε, υλοποιηθεί στην πράξη. Δεύτερον, για τις εξασφαλίσεις, τη μεταχείριση πιστωτών, συνέχεια της αξίας Νομίζουμε και εμείς, όπως και άλλοι, ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό το στοιχείο. Αν, υπάρχει, αν υπάρχουν ε, περιουσιακά στοιχεία που απομένουν σε έναν αντισυμβαλόμενο, θα πρέπει αυτοί να μετρούνται ε, με το σωστό τρόπο. Δημόσιες αρχές. Ε, η Κομισιόν υποστηρίζει όλες τις σχετικές τροπολογίες. Έχουμε όμως να κάνουμε μία παρατήρηση, την οποία κάναμε και όταν συζητήσαμε την έκθεση των εισηγητών. Η αρχιτεκτονική επιπτία. Ε, το ενιαίο, η ενιαία αρχή ε, εξυγίανσης ε, όταν συζητήσαμε εκείνο το θέμα ε, είχαμε πει ότι σε καιρό ειρήνης είναι εύκολο να συμφωνήσουμε σε αυτά τα θέματα. Ε, ε δεν ξέρουμε αν το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση ε, κρίσης. Ίσως ενδεχομένως λοιπόν πρέπει να, υπάρχει, να προβλέπεται και μια ρήτρα αναθεώρησης, να μην εγκαταλείψουμε εντελώς, εντελώς αυτή την ε, ιδέα, αυτή την προσέγγιση, αλλά να υπάρχει και η δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε στις καταστάσεις. Ευχαριστώ, Βάτρικ. Να ξαναδώσω το λόγο στους συνεισηγητές με την ίδια σειρά, ε, αντίθετη σειρά Γιάκοπ, συμφωνείς και εσύ. Παρακαλώ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Να τονίσω ότι ορισμένες από τις πιο τολμηρές τροπολογίες που υποβάλαμε ως μεμονωμένοι βουλευτές Ίσως ορισμένες θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο κείμενο τώρα και ορισμένες άλλες θα μπορούσαν ε, να μας βοηθήσουν ε, στη συζήτηση άλλων τμήματων του πακέτου ΕΜΙΡ. Νομίζω ότι ο Πάτρικ και οι συνεργάτες του διατύπωσαν πολύ σωστά το πακέτο, αλλά η σειρά η αλληλουχία με την οποία παρουσιάστηκαν τα διάφορα, τα διάφορα τμήματα του πακέτου δεν ξέρω αν ήταν η καλύτερη. Θεωρώ ότι οι αναθεωρήσει του μηχανισμού υποπτίας θα έπρεπε να συζητηθούν πριν από την αναθεώρηση του μηχανισμού ανάκαψης και εξυγίανση. Αλλά τι να κάνουμε, θα επιχειρήσουμε να αντιμετωπίσουμε τι δυσχέρειε όσο καλύτερα γίνεται. Ξέρω ότι δεν έγινε επειδή θέλατε να μα δυσχεράνετε που το κάνατε αυτό, είχατε λόγου. θα αντιμετωπίσουμε όσο καλύτερα μπορούμε την κατάσταση και σίγουρα μια ρωμαλαία ε, ρήτρα αναθεώρησης θα μας βοηθήσει. Πιστεύω ότι πρέπει να επιχειρήσουμε να πάμε όσο πιο μακρύτερα μπορούμε σε αυτή τη φάση. Γιατί αλλιώ ε, θα χάσουμε μια σημαντική ευκαιρία. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε. Και μάλιστα χωρίς ε, αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η ΚΕΙ. Ναι. Νομίζω ότι θα είναι δύσκολο να τα περάσουμε όλα αυτά μαζί, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Υπάρχει, νομίζω, συνένεση από αυτών των τροπολογιών και υπάρχουν πολλοί τομείς ε, που μπορούμε να προωθήσουμε. Αλλά ένα σημείο επί του οποίου ε, διαφωνώ α, εδώ και πολύ καιρό με τον Ιάκομπ είναι το τελευταίο τμήμα του προγράμματος αυτό. Έχουμε δουλέψει εδώ και πολύ καιρό για το Έμιρα δεν είναι κάτι που προέκυψε τώρα τελευταία, δεν συνδέεται με όλα τα άλλα. Εντάξει, ίσως είναι λυπηρό τώρα που δεν έγινε νωρίτερα, αλλά επειδή είναι τεχνικό το θέμα, πρέπει να ε, εγκρίνουμε ένα σαφές κείμενο, αλλά να αφήσουμε και ανοιχτή οποιαδήποτε δυνατότητα και άλλων ευρωπαϊκών μηχανισμών ε, να μπορούν να ε, ενταχθούν σε αυτό το πακέτο. Θέλω λοιπόν αυτό το θέμα να καταλήξει τάχιστα γιατί θέλουμε να υπάρχει και νομική βεβαιότητα. Όσο νωρίτερα λοιπόν τόσο καλύτερα. Αυτό ε, ε, το τμήμα έπρεπε βέβαια να αρχίσει να ισχύει αμέσως μετά το ΕΜΙΡ. Θέλω λοιπόν να το ξεχωρίσω από την ευρύτερη συζήτηση υποπτίας. Αλλά επειδή έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ και σε πολλά άλλα θέματα, Ελπίζω να εγκριθεί και αυτό σύντομα και όλες τις επόμενες συζητήσεις που σίγουρα θα μας απασχολήσουν ε, πάρα πολύ για το ε, υπόλοιπο τμήμα του θέματος ε, θα συνεχιστούν. Αλλά αυτό θέλω να περάσει γρήγορα. Ευχαριστώ και η ψηφοφορία ανάλογα με τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων αλλά από ό,τι κατάλαβα θεωρούν ότι οι συνεισηγητές ότι θα τα πάμε καλά. Η ψηφοφορία λοιπόν θα είναι στην Επιτροπή μας 24-25 Ιανουαρίου και αργότερα στο Ολομέλεια. Φυσικά θα γίνει και συζήτηση. Ψήφισα για την... Ε, συγγνώμη, μίλησα για την ψηφοφορία στην Επιτροπή. Όχι, όχι, οι κανόνες μας είναι σαφείς. Τους ξέρετε, πριν ψηφίσουμε πάντα κάνουμε ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή. Αλλά σας ευχαριστώ που μου το θυμήσατε. Υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν βλέπω να έχει κανείς τίποτα άλλο. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει την επόμενη Δευτέρα 3 με 6. Λήξη της συνεδρίας. Ευχαριστώ πολύ.